και έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά από την 27η Οκτωβρίου. Δεν βλέπω σχόλια, συνεπώς εγκρίνονται. Έχω ορισμένες ε, πληροφορίες να σας δώσω την περασμένη.